θα δώσει όθηση στην περιφερειακή ολοκλήρωση οπότε θα έχει άμεσα αποτελέσματα στη ζωή των ε, κατοίκων και αυτό είναι πάντα θετικό για τους πολίτες μας γι' αυτό και ψήψα υπέρ Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασμάρικ Ο κύριος Πόσελτ έχει το λόγο για ένα λεπτό Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τη στρατηγική του Δούναβη ως κάτι το βαθύτατα ευρωπαϊκό. Συνδέει την Γερμανία που ήταν ιδρυτική χώρα με νεότερες χώρες όπως τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, την επόμενη υποψήφια χώρα δηλαδή την Κροατία με μια χώρα που προσπαθεί να γίνει υποψήφια, τη Σερβία και χαίρομαι για το ότι συμπεριλαμβάνει την Τσεχία και το Μαυροβούνιο και κάποιες άλλες χώρες που ανήκουν ιστορικά στην Ευρώπη και συνδέονται με τον Δονοβή. αλλά μην ξεχνάμε και τη Βαβαρία. Εάν ήταν ανεξάρτητη, θα ήταν μετά τη Ρουμανία το δεύτερο μεγαλύτερο κράτος που θα βρεχόταν από τον Δούναβη. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόθεση της στρατηγικής του Δούναβη. Grazie collega, ora diamo la Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντάνιελ Ανάνε για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε και πάλι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει βάρος στην εμφάνιση και όχι στην ουσία. Το κίνητρο και όχι το αποτέλεσμα. Ψηφίσαμε εδώ πέρα ψηφίσματα που καταδικάζουν την Κίνα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πραγματικό κόσμο. Απομονώνει την Ταϊβάν, συμφωνήσαμε να απολύσουμε όπλα στο κομμουνιστικό καθεστώς του Πεκίνου, συνεργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εναλλακτικό του GPS, το οποίο το λέει τεχνολογικό υπεριαλισμό ο πρόεδρος Σαρκοζή. Βλέπετε πως η υποκρισία εδώ πέρα είναι η βασική μας αρχή. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά χρηματοδοτούμε τη Χαμάς, δεν μιλάμε τους αντιφρονούντες ε, που είναι κατά του Κάστρο εντό των συνόρων μα ε, όταν πάνε στραβά τα νομοψηφίσματα τα αγνοούμε και πάλι λέμε ότι εμεί είμαστε καλοί. Και τώρα θα έχουμε το εκπληκτικό θέαμα του να στέλνουμε τη Βαρόνη Άστον ω εκπρόσωπο για τα εξωτερικά στην Κούβα και στο Ιράν να του πει ότι δεν είναι δημοκρατικέ χώρε. Που αυτή δεν έχει εκλεγεί ποτέ. και δεν έχει εκτεθεί ποτέ στην κρίση των συμπολιτών της. Να ευχαριστήσω τέλος τους πολίτες της Μασαχουσέτης που ξεκίνησαν την επανάσταση και ε, είναι κατά της ιδέας του ότι μπορούν να επιβάλλονται φόροι χωρίς να τους θέλει ο λαός. Πρέπει να ξεκινήσει. Mezzo minuto in più, cioè un terzo di quello che era in più di quanto avrebbe dovuto. Onorevole Piotrowski. Α, ναι. Σας έδωσε περισσότερο χρόνο από αυτόν που είχατε. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριο Ποτρόφσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να εκφράσω την απόψή μου για το ότι περάσαμε ψήφισμα για τις επιθέσεις κατά χριστιανικών μειονοτήτων. Οι ευρωβουλευτές είναι εξοργισμένοι από τις επιθέσεις σε χριστιανικές μειονότητες γιατί επιτιθέμεθα έτσι στη βάση των Ευρωπαϊκών Εθνών. Εάν θέλουμε να είμαστε πίστευτοι, θα έπρεπε να είχαμε δεχτεί τις δύο τροπολογίες ε, της ε, ομάδας μας ε, που μας αποστασιοποιούν από την απόφαση του ΕΔΑΔ για τους σταυρούς της αίθουσας διδασκαλίας. Λοιπόν, που δεν συνέβη αυτό γιατί πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικός είναι ο χριστιανισμός για την ιστορία και τον πολιτισμό μας και να προωθούμε και να προστατεύουμε αυτές τις αρχές και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε, σου έδωσα το λόγο παρότι δεν είχες δικαίωμα γιατί οι γραπτές, οι, ε, ε, συγγνώμη, οι προφορικές επεξηγήσεις αφορούσαν μονάχα τη στρατηγική για το Δούναβι. Εν πάση περιπτώσει ε, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει επεξήγηση ψήφου επί των ε, κατεπηγόντων και αυτό το λέω και για τις μελλοντικές συζητήσεις μας. Επαναλαμβάνω ότι μονάχα σχετικά με την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον, για τον Δούναβη μπορείτε να πάρετε το λόγο για επεξήγηση ψήφου. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω για τις διακρίσεις εις βάρος των χριστιανών στην Αφρική και την Ασία, αλλά βεβαίως θα μιλήσω τώρα για το Δούναβι. Ή ε, για κάτι. Ναι, για τον Σημαντικός, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός στην Ευρώπη, μικρότερος μόνο από τον Βόλγα. Διατρέχει δέκα ευρωπαϊκές χώρες Γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την περιοχή, γιατί η περιοχή του Δούναβη έχει χώρες που είναι σε κρίση και κράτη μέλη της Ένωσης. Οπότε πρέπει να υπάρχει κάποια αλληλεγγύη από μέρος μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ζιμπράσκη και ολοκληρώνουμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για τον Δούναβη. Γιατί βεβαίως γινόμαστε έτσι πιο ανοιχτοί προς κάποιες περιοχές που έχουν κάτι το κοινό. Όπως παραδείγματος χάρη οι χώρες που ενώνει αυτός ο ποταμός. Χαίρομαι επίσης για τις ε, τροπολογίες ε, των Ευρωπαίων, για το ότι οι Ευρωπαίες, ε, με συγχωρείτε, οι τροπολογίες των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών δεν συμπεριλήφθησαν τελικά. Θα ήθελα τώρα και άλλες περιοχές να αποτελέσουν αντικείμενο της προσοχής μας, ίσως και η περιοχή του Όντερ. Ευχαριστώ κύριε και ο κύριος Ματζάρος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω κάποια πράγματα για την Κίνα ακόμα. Γιατί ψήφισα υπέρ. Ε, όχι, δεν γίνεται. Εξήγησα ήδη ότι δεν είναι δυνατόν να κάνετε επεξηγήσεις ψήφου επί των κατυπηγόντων. Μπορείτε να μιλήσετε μονάχα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Δούναβη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι η ε, διαδικασία. Ωραία. Επομένως δεν θέλετε να μιλήσετε. Άλλες ε, παρεμβάσεις. Τα πρακτικά της παρούς συνεδριάσεως θα υποβληθούν ή στην, ε, για, έγκριση στο Κοινοβούλιο την επόμενη ε, ολομέλεια και όλα τα ψηφίσματα θα αποσταλούν στους αποδέκτες τους. Επομένως, λύγεται η συνεδρίαση.